οι εν λόγω ορισμοί θα δημοσιευθούν στα πρακτικά αυτής τη συνόδου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μέχρι την έγκριση των πρακτικών, οι ορισμοί πρόκειται να θεωρηθούν ως εγκριθέντες.